Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας και επαναρχόμαστε στις ψηφοφορίες. Είχαμε προχωρήσει χθες αρκετά γρήγορα όλοι. Προσπαθήσαμε γι' αυτό και τα καταφέραμε. Συνεχίζουμε λοιπόν και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό θα έχουμε ολοκληρώσει μέσα στο πρωινό της εργασίας μας, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει σήμερα το απόγευμα να είμαστε ελεύθεροι για να ασχοληθούμε με άλλες δραστηριότητες δημοσιονομικού βέβαια χαρακτήρα ή άλλου. Αυτά. Υπάρχουν κάποια λαθάκια στη χθεσινή ψηφοφορία που πρέπει να τα διορθώσουμε. Ο εισηγητή θα μας τα εξηγήσει αυτά. Και μετά, σύμφωνα με τόσα αποφασίσαμε χτες, θα ψηφίσουμε σήμερα την κατηγορία 5 για τα άλλα όργανα, έκθεση Derek Von, και μετά θα ψηφίσουμε ακόμα το 1α, 1β και την κατηγορία 4. Και θα τελειώσουμε με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προετοιμασίες. Λοιπόν, κύριε Σιγητά, έχετε να μας δώσετε κάποια διευκρίνηση, έτσι δεν είναι, για την χθεσινή ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ψηφίσαμε χθε ε, για τον τομέα 3β σχετικά με τρεις γραμμές, Youth in Action, Info Outlet και το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, ψηφίσαμε ένα εκατομμύριο στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές. Εμείς θέλαμε ένα εκατομμύριο πάνω από το, το σχέδιο προϋπολογισμού ενώ εχθές είπαμε ότι ήταν ένα εκατομμύριο πάνω από αυτό την πρόταση του Συμβουλίου. Λοιπόν, συμφωνούν οι συνάδελφοι να είμαστε πάνω από το σχέδιο του προϋπολογισμού ένα εκατομμύριο. Δηλαδή και σε αυτήν τη γραμμή και στις άλλες γραμμές αν υπάρχουν λάθη θα ισχύσει η συμφωνία που κάναμε στους συντονιστές. Καλώς. Ε, νεολαία στη δράση, Fashion Outlet και Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013. Είναι αυτές οι τρεις γραμμές. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει παρεξήγηση από αυτόν. Διότι χτες υπήρξε κάποια σύγχυση όταν ψηφίσαμε. Γενικά μιλώντας, για διάφορες γραμμές υπήρξε συμφωνία μεταξύ των συντονιστών εδώ και δύο μέρες, ώστε να πάμε πέρα από τα ποσά του σχεδίου προπολογισμού. Αυτό θα το δούμε και σήμερα για ορισμένες γραμμές στην κατηγορία 1α και στην κατηγορία 4. Και αυτό ίσχυε και για τις τρεις γραμμές της κατηγορίας 3β που ψηφίσαμε χτες. Λοιπόν, για το 3β το ξεκαθαρίσαμε και θα ψηφίσουμε τώρα τις άλλες κατηγορίες. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Συνεπώς, έχετε όλοι τις ε, κάρτες για την ψηφοφορία, έτσι. Η ομάδα μου πρέπει να μου πει, δεν μπορώ να ψηφίσω ή μπορώ να ψηφίσω. Οπότε μου λένε ναι, μπορώ να ψηφίζω. Γιατί οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ φαίνεται ότι αργούν να ξυπνήσουν και δεν είναι εδώ ακόμα. Συνεπώς, other sections, άλλα τμήματα. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας όλοι. Λοιπόν, αρχίζουμε με τα θεμέλια της εργασίας μας, που είναι και το αποτέλεσμα της συμφωνίας που είχαμε στη συνδιαλλαγή με το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεκινάμε δηλαδή με τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Και όλες οι τροπολογίες έχουν υποβληθεί από τον δικό μας τον εισηγητή με τη συμφωνία των συντονιστών εκ μέρους του Προεδρείου. Αυτή είναι η σχέση που έχουμε τώρα με το Προεδρείο και προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ καρποφόρα. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε μαζί τον πρώτο πίνακα, όλο μαζί, αλλά υπάρχει προφορική τροπολογία για τον Νίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ο εισηγητής μας θα μας εξηγήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι τροπολογίες στη σελίδα 2 που έχουν μπροστά τους οι συνάδελφοι αντικατοπτρίζει την συμφωνία που πετύχαμε στη συνδιαλλαγή. 1,9% που περιλαμβάνει το κόστος και για την Κροατία. Στο κείμενο όμως δεν γίνεται μνήα στον νίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας πέρα από τη συμφωνία που είχαμε στη συνδιαλλαγή που ήταν να μειώσουμε το ποσό που πάει στον ε, οίκο αυτό του χρόνου κατά 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η προφορική τροπολογία λέει ότι ε, τη γραμμή 3247 μετά βάσει τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στη συνδιαλλαγή. Καλώς. Εντάξει, είναι σαφές για όλους. Συνεπώς, από εδώ και πέρα προτείνω να ψηφίσουμε όλη τη σελίδα. Όλα μαζί όσα αναφέρονται στη σελίδα αυτή και τις τροπολογίες επί του κειμένου. Γιατί αυτή είναι η συμφωνία που πετύχαμε στη συνδιαλλαγή. Συνεπώς, το σύνολο των τροπολογιών στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου, όλες μαζί, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Καμία. Ευχαριστώ. Α, υπάρχει μία. Ο Τζέιμς. Ωραία. Θα το σημειώσουμε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για το δύσκολο έργο του. Τώρα, Έχουμε κάποιες άλλες τροπολογίες που πρέπει να τις ψηφίσουμε χωριστά. Πρώτα απ' όλα, τροπολογία εκ μέρους του Προεδρείου που έχει να κάνει με μια τεχνική διευκρίνηση η οποία καθίσταται αναγκαία εξαιτία του δημοσιονομικού κανονισμού. Παρακαλώ κύριε Σιγητά, εξηγήστε μας την τεχνική φύσεως αυτή η τροπολογία. Νομίζω ότι συνοψίσατε καλά, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια τεχνική φύσεως τροπολογία που αντικατοπτρίζει τα όσα αναφέρονται στο δημοσιονομικό κανονισμό και κυρίως μιλάει για τα κονδύλια για τα κτίρια που είναι εξωτερικά έσοδα, είναι μια μεταφορά. Τεχνική τροπολογία που μπορούν να στηρίξουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε. Υποθέτω να υπάρχει πρόβλημα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Μία. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα επίσης, η επόμενη. Έχει αποσυρθεί. Πρέπει όμως να ψηφίσουμε τις δύο τροπολογίες, οι τρεις, Για εξηγήστε μας τις τρεις τροπολογίες που πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στη σελίδα 2 βλέπετε ότι υπάρχουν τρεις τροπολογίες που πρέπει να ψηφίσουμε και που έχουν να κάνουν με το κείμενο. Η πρώτη είναι του ECR, η οποία αναφέρεται στην διαφάνεια και την λογοδοσία που έχει να κάνει με τις γενικές δαπάνες. Η δεύτερη είναι στην 3428 και έχει να κάνει 3248 και έχει να κάνει με το κάτω από 1000 ευρώ για ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με την Ανατολική Ευρώπη. Πολλοί από εμά θα πούνε ναι, ναι, αλλά ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα, οπότε να την καταψηφίσουμε. Και όσον αφορά την τρίτη τώρα, που ήταν για 200.000. Η τρίτη έρχεται από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την ΑΦΚΟ, και λέει ότι μέχρι τις επόμενες εκλογέ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δαπανηθούν κάποια χρήματα για μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να δώσουν μεγαλύτερη δημοσιότητα στις ευρωεκλογέ αυτές. Αυτό βέβαια δημιουργεί κάποια προβλήματα στην δίκηση και μπορεί να μην θέλουν γιατί αντιτίθεται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό είναι το ένα επιχείρημα. Και το άλλο του επιχείρημα είναι ότι θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Πώ θα αποφασίσουμε ποιο θα πάρει τα χρήματα και πώ θα δαπανηθούν. Γι' αυτό και προτείνω να την καταψηφίσουμε και αυτή. Συνεπώ, για τι τρει προτείνω να τι καταψηφίσουμε. Και τι τρει λοιπόν. Unblock Όλες μαζί και τις τρεις. Α, όχι βλέπω. Η άλλη δεν διαφωνεί. Πρώτη τροπολογία. Η 553. Ο εισηγητής διαφωνεί. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Του κυρίου Σόνιξ τώρα η τροπολογία. Διαφωνεί ο συγκητής. Υπέρ παρακαλώ. Το Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Της ε, Σταγματικής Επιτροπής. Διαφωνεί ο συγκητής. Υπέρ παρακαλώ. Η άλλη που έχει συνεπογράψει. Κατά. Οι υπόλοιποι. Αποχές. Απορρίπτονται. Και οι τρεις λοιπόν με διαφορετικές όμως πλειοψηφίες μεταξύ τους. Ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Τελειώσαμε με το Κοινοβούλιο. Περνάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Αυτά για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στη συνέχεια. Ελεκτικό συνέδριο. Μαζί της δύο τροπολογίες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Για τον διαμεσολαβητή. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Κύριε Σίγητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. είναι μια θέση που προβλέπεται για στήριξη του Ombudsman, ο οποίος λέει ότι πρέπει να έχει ένα νέο λογιστή που να τον ορίσει ο ίδιος. Αυτό λέει η τροπολογία. Μία θέση δηλαδή για λογιστή όσον αφορά τον Ombudsman. Δεν υπάρχει πρόβλημα από αυτού. Καλώς, είναι προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε, συνεπώς, όλες τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με το διαμεσολαβητή και αυτήν. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για τον επόπτη προσωπικών δεδομένων τώρα. Πάλι όλες μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τώρα. Μαζί οι τροπολογίε υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, εγκρίνονται. Επιτροπή των Περιφερειών, μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται επίσης με την ίδια πλειοψηφία. Γυρίζουμε σελίδα. Υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Η Γκουε διαφωνεί. Αποχή. Α, αποχή. Τρεις κατά και μία αποχή. Υπάρχει κατά τμήματα για την 572 εισήγητης, παρακαλώ. Κατά. Υπέρ είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 462. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Πράσινη και ECR. Και η Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη συνέχεια έχουμε ένα κατάλογο τροπολογιών που έχουν αποσυρθεί. Συνεπώς, για τα άλλα όργανα τελειώσαμε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Οπότε, τώρα ερχόμαστε στην κατηγορία 1α. Θέλετε το λόγο κύριε Σιγητά. Παρακαλώ. Παρουσιάστε μας την ψηφοφορία για το 1α. Για τον τομέα 1α αποφασίσαμε στη συνεδρίαση των συντονιστών να ζητήσουμε ευελιξία για ένα συνολικό ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας είναι πιθανό να έχουμε κάποια περαιτέρω περικοπή σχετικά με αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει στις διάφορες γραμμές. Εγώ λέω για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε κατά τη διαδικασία αυτό το ποσό Για να κρατήσουμε λοιπόν αυτήν την ευελιξία θα έλεγα για την διαβίου μάθηση να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό έναντι του σχεδίου προϋπολογισμού. Καταλάβατε όλοι αυτή την πρόταση. Πολύ ωραία. Αρχίζουμε αμπλοκ με τον συμβιβασμό, μόνο για τους αριθμούς. Πρώτος υποτομέας για τις γραμμές που θέλουμε να ξεπεράσουμε το σχέδιο του προπολογισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερος υποτομέας που θέλει να αποκαταστήσει το αρχικό σχέδιο υπέρ. Αποχές μία. Εγκρίνεται. Τρίτο. Στον πίνακα τρία στο παράρτημα. Ποιος είναι υπέρ. Αποχές. Ευχαριστώ. Τώρα, χωριστή ψηφοφορία όσων δεν καλύπτονται από, τις, από το συμβιβασμό. Ο 700, η 706 τροπολογία είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Της τροπολογίας της Γκουε. Α, η κυρία Αντράσεν. Κατά αποχές απορρίπτονται αυτές οι τροπολογίες Οι 993 των πρασίνων είναι κατά ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές Έχουμε και άλλες τροπολογίες της ΓΚΟΥ 600 κατά ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41-39 της κυρίας Βέρτμαν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 της ΕΚΟΝ υπέρ. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 695 της ΓΟΥ είναι κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ECR 599 είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4487 είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τρεις τροπολογίες. 8,78 και άλλες δύο που είναι ταυτόσιμες. Είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά η ίδια πλειοψηφία. 351 είναι υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη γραμμή. 677 της Γκουε είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 964 ε, των πρασίνων κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4166 της κυρίας Βέρτμαν είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται με, την με τον ίδιο συσχετισμό. Επόμενη γραμμή, ΙΜΚΟ 541, με μια προφορική τροπολογία του εισηγητή μας. Ο εισηγητής ζητά να ψηφιστεί 1,5 εκατομμύριο αποθεματικό. Α, ένα λεπτό, ένα λεπτό. 1,5, 1,5. 1,5 εκατομμύριο ευρώ να μπουν στο αποθεματικό. Υπό όρους, όπως τις έχετε στην προφορική τροπολογία. Αν θέλετε να σας τη διαβάσω. Όλοι την έχουν μπροστά τους. Όλοι έχουν μπροστά τους τους όρους. Υπέρ αυτής της ε, πρότασης με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά κανείς αποχές ομόφωνα. Είναι παρούσα η Κομισιόν και ενημερώνεται για αυτήν την ψηφοφορία σχετικά με τους όρους για την άρση του αποθεματικού. 8077 της κυρίας Γκρέσλερ. Έχει καταπέσει. Η εξαφανίστηκε. Ωραία. Στα σχόλια τώρα. 7.42 είναι υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άντε 743 είναι κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Αρχίζει ψηφοφορία. Έχω και εδώ μηχανάκι. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Είσαι υπέρ ή κατά, Ρίτσαρτ. Κατά. Άλντα, είσαι υπέρ. Ωραία, άρα εξουδετερώνει το ένα στον άλλο. 18-15 ή 19-16 όπως θέλετε. Πλειοψηφία υπέρ. Αλλάξτε θέση άμα έχετε πρόβλημα. Αλλά αν εξουδετερώνει το ένα στον άλλο συστηματικά, μπορείτε να μείνετε εκεί που είστε. 42-55 του κύριου Ντάρντεν είναι υπέρ, εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 620 της Γκουε είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 387 των μεταφορών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 673 της Γκουε είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 4161 της κυρίας Βέρτμαν για την, για την επιληψία. Είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Εφτά σαραντατέσσερα της Άλντε για εταιρική σχέση στο νερό. Διασκεδαστικό λέει ο πρόεδρος, δεν του αρέσει πίση, γιατί υπέρ. Για να δούμε λοιπόν ηλεκτρονικά. έχουμε έναν σοσιαλιστή παραπάνω στην πισίνα. Ένα σοσιαλιστής λοιπόν μπορεί να πέχει. Πέρας της ψηφοφορίας. 18-18 απορρίπτεται. Είναι μυστική ψηφοφορία, δεν ξέρουμε ποιος ψήφισε τι. 773 της Άλντε, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 774 της Άλντε είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έχουμε πλειοψηφία κατά. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Για την 774. Innovative Products and Services. Ψηφίστε κόσμο, λέει ο πρόεδρος. Πέρα της ψηφοφορίας. 17-18. Απορρίπτεται. 9.65 των πρασίνων. Είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 966 των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1048 της ΙΜΚΟ για την αλλαγή ενός τίτλου είναι υπέρ ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 της Επιτροπής Πολιτισμού είναι υπέρ ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε σελίδα. 899. Support Brain Trust. Έχει καταπέσει. Λοιπόν, δεν έχει Brain Trust, λέει ο πρόεδρος. 43-41 του κυρίου, της κυρίας Γκιόγκς. Είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42.50 του κυρίου Γκάιερ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 550. Είναι υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. κατά. Επαλήθευση 550 του, το, του ΕΦΔ. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ 13 κατά, 2 αποχές, εγκρίνεται. Αποθεματικά. χωριστή ψηφοφορία εδώ. Ένα πρώτο τμήμα, ένα ποσό από 1,5 εκατομμύριο που δίνεται στην οθόρυτη. Υπέρ ο εισηγητής, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, third authority μέχρι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Κυρία Ανδρέας. Εγκρίνεται. Και η άλλη τροπολογία έχει αποσύρθει. Τελειώσαμε με το 1α. Bien, alors, nous allons prendre le 1. Πάμε στο 1β. Πριν ψηφίσουμε το 1β, προτείνω να πάμε λίγο πίσω και να πάμε σε αυτό που αναρωτηθήκαμε χτες για το με ποιο τρόπο δηλαδή πρέπει να διατυπώσουμε τα άτομα εκείνα τα οποία ανήκουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα της Κύπρου. Οι σοσιαλιστές μας μοίρασαν ένα χαρτί στο οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, προτείνουν μία λύση. Δεν ξέρω κατά πόσο πολιτικά είναι τέλεια, είναι κομψή πάντως. Capacity building προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση της κοινωνίας των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεκτημένο της και προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα για την εφαρμογή και τη χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το λόγο θέλετε, Φέραν. Ναι, ναι, θέλω να εξηγήσω τι εννοούμε δηλαδή πώς ονομάζουμε τελικά την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Υπάρχει και στον τίτλο των γραμμών του προπολογισμού, οπότε δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε και γι' αυτό το διαγράψαμε εντελώ από το κείμενο. Οπότε είναι πιο ουδέτερο το κείμενο αυτό και ρωτήσαμε και τις πολιτικές ομάδες και από ό,τι φαίνεται όλοι συμφωνούν. Ωραία, πολύ κομψό. Οι ναυτικοί λένε ότι κάποια στιγμή πρέπει να δώσουμε όσο γίνεται λιγότερες ευκαιρίες στον άνεμο. Συνεπώς, ποιος είναι υπέρ της διατύπωση αυτής. Κατά αποχές. Συνεπώς εγκρίνουμε τη διατύπωση αυτή που προτάθηκε. Δεν έχει να κάνει με τα ποσά, ε, δεν επανερχόμαστε στα ποσά ή στο στόχο της οικονομικής αυτής ε, στήριξης, πρόκειται για τη διατύπωση μόνο. Ωραία. Έτσι. Τώρα ερχόμαστε στο 1β. Σελίδα 71 μου λένε. Κάτω-κάτω στη σελίδα. Αρχίζει με τις διοικητικές δαπάνες. Θέλετε να μας τα παρουσιάσετε κύριε Σίγητα μήπως. Νομίζω, Πρόεδρε, για να συντομεύσουμε την ψηφοφορία σχετικά με το σχέδιο, σχέδιο δηλαδή την αποκατάσταση του αρχικού σχεδίου προπολογισμού, μπορούμε να ψηφίσουμε unblock, εκτός από τη γραμμή για την τεχνική βοήθεια στις περιοχές της Βαλτικής θάλασσας. Μπορούμε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα να τα ψηφίσουμε unblock, εκτός από αυτό. Ε, Η γραμματεία μου λέει ότι ε, εδώ υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος ότι επειδή δεν έχουμε προετοιμάσει με αυτόν τον τρόπο την ψηφοφορία πιθανόν να μας ξεφύγει κάποια γραμμή. Συνεπώς, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πρώτον να ψηφίσουμε συνολικά, όπως προτείνει ο εισηγητής, για να δούμε κατά πόσο υπάρχει πλειοψηφία, ώστε να καταλάβουμε ότι κάθε φορά που προτείνεται η αποκατάσταση του σχεδίου προπολογισμού συμφωνούμε ότι υπάρχει πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, υπέρ. Και μετά θα διαβάσουμε τις γραμμές μαζί και θα διασφαλίσουμε μαζί ότι δεν θα έχουμε ξεχάσει καμία γραμμή. Συμφωνείτε? Ωραία. Συνεπώς, επί της αρχής, ότι κάθε φορά που ο εισηγητής προτείνει να επανέλθουμε στα ποσά του σχεδίου προϋπολογισμού, συμφωνούμε. Επαληθεύουμε ότι υπάρχει πλειοψηφία από αυτού. Υπέρ. Κατά. Τέσσερις αποχές. Καλώς. Τώρα, από εδώ και πέρα. Θα πάω αργά-αργά για να μην ξεχάσουμε τίποτα. Στο τέλος της σελίδα 71, λέει ο πρόεδρος, χτες το κοιτάξαμε αυτό λίγο, πρόκειται για διοικητικές δαπάνες. Ολοκλήρωση του Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Ταμείου, δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Στην επόμενη σελίδα, όχι. ESF σύγκληση. Α, ναι, ναι, ναι, εδώ. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Λοιπόν, convergence, σύγκληση. Εδώ δεν υπάρχει αποκατάσταση σχεδίου προπολογισμού, συνεπώ πρέπει να ψηφίσουμε την 730 της Γκουίπερ. Διαφωνεί ο συγκεκριτής. Κατά. Άλντα, είσαι υπέρ ή κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45-17 είναι ίδια. Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Είμαστε υπέρ της αποκατάστασης, 350 δηλαδή, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια. Και ο εισηγητή διαφωνεί. Υπέρ παρακαλώ. Θέλεις το λόγο, Άλντα. Ναι. Εδώ έχουμε πάνω από το σχέδιο προπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση 602 και 500 Ναι, λέει ο πρόεδρος, αλλά στη γενική ψηφοφορία αποφασίσαμε ότι για όλες τις γραμμές όπου ο εισηγητής προτείνει να αποκαταστήσουμε το σχέδιο προπολογισμού, τα ποσά δηλαδή αυτά, αυτό ψηφίζουμε. Οπότε για την γραμμή αυτή, αυτό σημαίνει ότι κρίνουμε την 350. Άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τις υπόλοιπες, αυτή είναι η αρχή. Από την άλλη όμως η ψηφοφορία αυτή αναφέρεται στα ποσά μόνο. Συνεπώς κάθε φορά που υπάρχουν τροπολογίε επί των σχολείων, τότε ναι, πρέπει να τις ψηφίσουμε τις τροπολογίε αυτές. Εντάξει τώρα. Ωραία. Για τα σχόλια του 4578. Ο εισηγητή διαφωνεί. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το επόμενο καλύπτεται. Μετά έχουμε δοκιμαστικά σχέδια. Θα είναι σελίδα 74 στο γαλλικό κείμενο προφανώς. ο πρόεδρος πρέπει να ψηφίσουμε τα σχόλια. Α, όχι, είναι αποθεματικό. Αποθεματικό του 765. Το ζητάει Άλντε. Ο εισηγητής διαφωνεί. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε με το Ιαντιέφ. 359 τροπολογία. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπήρξε μια τροπολογία για το αποθεματικό που όμως αποσύρθηκε. Οπότε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη, Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, το είδαμε. Ευρωπαϊκή Δαφική Συνεργασία τώρα. Σελίδα 92 στο ελληνικό κείμενο. Έχει αποσυρθεί η σοσιαλιστική τροπολογία, οπότε αποκαθιστούμε με την 360 το σχέδιο προπολογισμού. Σωστά. Παρακολουθείτε όλοι. Γυρνάμε σελίδα. Στην ε, Επόμενη σελίδα. Για την ε, επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια δεν υπάρχει πια, έχει φύγει η εσωτερική τροπολογία, παραμένει 361 για την αποκατάσταση. Τα υπόλοιπα είναι δοκιμαστικά σχέδια. Στη συνέχεια πρέπει να ψηφίσουμε την τεχνική βοήθεια και διάδοση πληροφοριών και λοιπά για τη Βαλτική Σελίδα 94 στο ελληνικό κείμενο. Εδώ δεν έχουμε τροπολογία για αποκατάσταση του σχεδίου, άρα πρέπει να ψηφίσουμε εδώ όλες τις τροπολογίες. 747 πρώτα. Άλντε. Διαφωνεί ο εισηγητής με τον Μπόιν. Υπέρ. Κατά. Εδώ πρέπει να παληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για το 747 της Άλντε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Υπάρχει ένας σοσιαλιστής παραπάνω. Για αφαιρέστε ένα σοσιαλιστή. Ωραία. Πέρα τη ψηφοφορία. 18 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. Για τα ποσά έχει διακανονιστεί, αλλά υπάρχουν σχόλια. Για το 342. Σωστά. Σχόλια της δικιάς μας Περιφερειακής Επιτροπής. Ο εισηγητής συμφωνεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συναπώς. κρατάμε το ποσό του 747 με τα σχόλια της 342 τροπολογίας. Συνεπώς, ελπίζω ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή. Ε? Προσοχή. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν προπαρασκευαστικές ενέργειες και στην επόμενη σελίδα μέχρι το Ταμείο Συνοχής. Οι σοσιαλιστές έχουν αποσύρει την επιφύλαξή του. Τροπολογία 363 τώρα, η οποία αποκαθιστά το σχέδιο προπολογισμού. Άρα το ποσό του 363 κρατάμε. Ταμείο συνοχή συνεχίζουμε. Και εδώ έχουμε την τροπολογία 364, η οποία αποκαθιστά το ποσό του σχεδίου προπολογισμού. Και στη συνέχεια πρέπει να ψηφίσουμε την 766 των φιλελεύθερων που θέλει αποθεματικό και μένει στην τροπολογία της αυτή. Ο εισηγητής διαφωνεί. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 748. Έχει αποσυρθεί. Των φιλελεύθερων πάντα. Και τελειώσαμε με το αναβήτα. Όλα αυτά πάνε πολύ γρήγορα. Συνεπώς, περνάμε στο 4. Non, le... on va tellement vite que j'ai oublié. Πάμε τόσο γρήγορα που ξέχασα ότι το 4 το ψηφίσαμε χτες. Οπότε περνάμε στα δοκιμαστικά σχέδια. Tout le monde a les, les tableaux. Alors... Έχετε όλοι τον πίνακα. Έχουμε δύο πίνακες έναν πίνακα με τα σχέδια, τα δοκιμαστικά σχέδια και τα ποσά και ένα πίνακα με τα σχόλια που εξηγούν το περιεχόμενο των ε, προπαρασκευαστικών ενεργειών και δοκιμαστικών δράσεων. Αντικείμενο μακρών ε, συζητήσεων και εργασιών από πλευρά των συντονιστών. Κύριε Σιγητά, προτείνατε να ψηφίσουμε όλα μαζί, ε? υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρει τα δοκιμαστικά σχέδια. Περιμένουμε λίγο ώστε να έχουν όλοι μπροστά τους τους πίνακες. Και στα μέλη της ομάδας σας, Λόρα, λέει ο πρόεδρος της ομάδας μας. Γιατί βλέπω ότι τα μοιράζετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εμείς είμαστε κοινοβούλιο. Ξεκινήστε από το κοινοβούλιο. Bien. Λοιπόν, το έχετε όλοι. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλο μαζί τα ποσά πρώτα και μετά τα σχόλια. Μαζί λοιπόν τα σχέδια και για τα δοκιμαστικά και για τις προβάσεις Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Σχόλια τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ωραία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να ψηφίσουμε. Συγχαρητήρια στους εισηγητές. Ωραία. Πριν τώρα κηρύξουμε τη λήξη των εργασιών μας. Βλέπετε πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα. Του χρόνου μισή μέρα να σκεφτούμε να προβλέψουμε μόνο. Θα μας φτάσει αφού πήγαμε τόσο γρήγορα αυτή τη φορά. Αλλά προσοχή, ε, είσαστε σίγουροι ότι θα κοστούν διάφορες ε, κατηγορίες από τη δίκηση. Θα τις αναλάβω εγώ, έτσι, θα αναλάβω εγώ την ευθύνη. ότι κρατήσαμε την αίθουσα για τόσες μέρες και ότι τελικά δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε σήμερα το απόγευμα. Αλλά τι να κάνουμε, καλύτερα να λειτουργούμε έτσι, αποτελεσματικά, παρά το αντίθετο, να χρειαζόμαστε παραπάνω μέρες για την ψηφοφορία. Αλλά πριν τελειώσουμε, ας προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα θέμα που ο Σαλβαδόρ θέλει να μας εξηγήσει. Μάλλον ο Σαλβαδόρε ζήτησε να του το εξηγήσουμε. Πρώτον, την επόμενη εβδομάδα έχουμε δύο κατηγορίες ψηφοφορίας πολύ σημαντικές και κάποιες άλλες λιγότερο σημαντικές. Πρώτον, όπως γίνεται κάθε χρόνο, 8 μέρες μετά την ψήφιση των τροπολογιών επί του σχεδίου προπολογισμού, έχουμε την έγκριση του ψηφίσματός μας. Και εδώ έχουμε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών που λύγει. Πότε? 8 μου λένε. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι. Ε? Γι' αυτό πολύ σύντομα θέλω την επιβεβαίωση. Για το ψήφισμα, ναι. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε και να συζητήσουμε το σχέδιο Interim Report για το MFF, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα ψηφίσουμε στις 11 του μηνός, προκειμένου να υπάρχει αρκετός χρόνος για τις ομάδες να εξετάσουν την προσωρινή αυτή έκθεση, η Επιτροπή Προπολογισμών δηλαδή, ενδεχομένω να υποβάλουμε τροπολογίε, ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στο Στρασβούργο στις 23 Οκτωβρίου. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προβλέψει μία έκτακτη κατά κάποιο τρόπο συνεδρίαση που προστίθεται το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου και η οποία θα αφοσιωθεί και θα αφιερωθεί στην συζήτηση της προσωρινής αυτής έκθεσης ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να προετοιμάσουμε την ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα στις 11 Οκτωβρίου. Προς το παρόν, έχουμε προβλέψει να χρησιμοποιήσουμε την δεκάτη και την ενδεκάτη του μηνός, πρωί και απόγευμα και τις δύο μέρες, για να ψηφίσουμε την προσωρινή αυτή έκθεση και το ψήφισμα. Και βέβαια την υπόλοιπη μερίσια διάταξη που προβλέπει κάποιες εκθέσεις επί των οποίων γνωμοδοτούμε. Στρέφομαι τώρα προς την γραμματεία δεν είμαι σίγουρος ότι χρειαζόμαστε πέντε μισές μέρες την επόμενη εβδομάδα. Ε? Πρέπει να δούμε. Καλώς. Προς το παρόν, βάλτε αυτές τις ημερομηνίες στην ατζέντα σας και αν τα καταφέρουμε, όπως αυτή την εβδομάδα, να εξοικονομήσουμε μισή μέρα ή παραπάνω, νομίζω ότι κανένας δεν θα στενοχωρηθεί. Κρατήστε λοιπόν αυτές τις ημερομηνίε. Μπορεί να γυρίσετε σπίτι σας με σήμερα νωρίτερα. Πάντως, μέχρι το τέλος του πρωινού θα σας επιβεβαιώσουμε ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για το ψήφισμα. Α, τώρα το ξέρω. Όντως, η 8η Οκτωβρίου είναι η προθεσμία, 12 το μεσημέρι και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει περάσει. Οπότε εδώ δεν έχουμε μεταφυσικού είδους προβλήματα, δεν χρειάζεται. Σαλβατόρε, εντάξει. Για μένα είναι απλώς το ότι πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις που θα ψηφίσουμε την 5η 11 του μηνός. Οπότε για τις προθεσμίες ήθελα εγώ να ξέρω. Μπορούμε μήπως να ψηφίσουμε στις 10 καλύτερα αντί για τις 11. Ξέρω ότι εξαρτάται από τις προθεσμίες και πώς η γραμματεία μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αίτημα. Αν γίνεται πάντως, αν κάποιες ψηφοφορίες τουλάχιστον μπορούμε να τις κάνουμε την Τετάρτη 10 του μηνός, θα ήταν προτιμότερο. Πρόεδρος, εφόσον ε, πολιτικά δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να ψηφίσουμε και στις 10 για το ψήφισμα. Ίσως και την ε, προσωρινή έκθεση, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα που έχουν οι συγητές μας να πετύχουν συμβιβασμούς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω και να πιέσω. Είναι πολύ δύσκολα ζητήματα αυτά μπορούμε να προσπαθήσουμε να θέσουμε ως στόχο, αν μη τι άλλο για το ψήφισμα, να ψηφίσουμε στις 10 του μηνός. Και ή δυνατόν και για το MFF. Ωραία, με Ροζαλούκ είναι εδώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κρατήστε στο κεφάλι σας ότι μάλλον το MFF, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα το ψηφίσουμε την Πέμπτη. Έλγα, σε πολλές ε, χώρες αυτό που αποσχολεί είναι ο προπολογισμό της Ευρωζώνης και πώς θα το πετύχουμε να βάλουμε ό,τι πρέπει εκεί. Τον Οκτώβριο πολλές ιδέες και πολλές ε, αλλαγές στις συνθήκες συζητιούνται και τι γίνεται εμείς συζητάμε τώρα με τον παλιωμοδίτικο τρόπο το, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενώ υπάρχουν νέε ιδέες στα κεφάλια των ηγετών μας. Οπότε τι θα γίνει τώρα με το Συμβούλιο και τη συνάντηση που θα έχουμε τον Οκτώβριο ή με το MFF. Ίσως αυτά τα οποία συζητιούνται τώρα να βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πολιτική κατάσταση και ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε ξανά. Ας ελέγξουμε τη μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, μπορεί να υπάρξουν νέε ιδέες που να πρέπει να τι λάβουμε υπόψη μα. Γι' αυτό λέω να ξανασυζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Πρόεδρος, σωστά, θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε κατά την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης, για το οποίο είμαι εγώ εισηγητής όσον αφορά την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής που κάνει η κυρία ε, Μάριαν Τάισεν που είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας για τις προτάσεις του Προέδρου Φαν Πάου προκειμένου να ενισχυθεί Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το Κοινοβούλιο, δηλαδή η ΕΚΟΝ, αμέσως από τον Ιούνιο ζήτησε, αμέσως μετά το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, να ετοιμάσει έκθεση πρωτοβουλίας και να ψηφιστεί τον Οκτώβριο, όταν θα γίνει το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή να ψηφίσουμε και εμεί στην Ολομέλεια. Οπότε, Χέλγα, ειλικρινά, εξεπλάγει και βρίσκω ανησυχητικό το ότι στο κείμενο το οποίο κυκλοφόρησε εδώ και 15 μέρες ο πρόεδρος Φαν Ρομπάι, σαν έναν οδηγό για τις διαπραγματεύσεις και σαν άτυπο ερωτηματολόγιο, προς τους ε, συναδέλφους του Συμβουλίου για να προετοιμαστεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Με εξέπληξε λοιπόν που μέσα λέει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και έναν κεντρικό προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη. Πριν από δύο μέρες είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο Φαν Ρομπάιου. Ε, δεν ήταν ακριβώς ε, τέτα τέτ, ήταν για ένα άλλο θέμα. Παρ' όλα αυτά προσπάθησα να καταλάβω καλύτερα τι, ποια είναι η ιδέα του. Όπως η Έλγα, όπως και άλλοι, έτσι και εγώ, έχω διαβάσει δηλώσεις από διάφορους ηγέτες επικεφαλής, δηλαδή και κυβερνήσεων. Και από ό,τι φαίνεται επικρατεί μεγάλη σύγχυση. Σίγουρα ο καθένας έχει στο μυαλό του διάφορα στοιχεία έτσι, στρατηγικής, τακτικής που θέλει να ακολουθήσει. Πάντως, υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις πίσω από την διατύπωση αυτή προπολογισμό της Ευρωζώνης. Η μία αντίληψη λέει ότι αν έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, δηλαδή ένα ταμείο που διευκολύνει τις χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, είναι δυνατόν να έχουμε αργότερα και ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων Τραπεζικών Καταθέσεων ή στήριξη των τραπεζών οι οποίες απειλούνται με πτώχευση. Ο πρόεδρος Μπαρόσο ανακοίνωσε ότι θα κάνει σχετικές ε, ανακοινώσεις. Συνεπώς πρέπει να βρεθεί μια οικονομική εγγύηση που θα καθησυχάζει τις αγορές και που θα δείξει ότι το ταμείο αυτό που θα δανείζει θα έχει ως βαθμολόγηση το τριπλό α. Οπότε πρέπει να δούμε ποιοι πόροι θα συμπεριληφθούν σε αυτό το ταμείο. Αυτή είναι μια πρώτη υπόθεση, ένα πρώτο μοντέλο, μια πρώτη αντίληψη. Ορισμένοι όμως αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτός ο προπολογισμός της Ευρωζώνης θα μπορούσε να έχει επίσης ως στόχο το να βοηθάει με οικονομική στήριξη, επιδοτήσεις κατά κάποιο τρόπο, χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πρόγραμμα βοήθειας. Άρα είναι σαν να ξαναφτιάχνουμε το Ταμείο Συνοχής ή τέλος πάντων να το συμπληρώνουμε για αυτές τις χώρες. Όλα αυτά όμως μέσα σε μεγάλη σύγχυση. Και προσθέτω, και αυτό είναι που με έκανε κυρίως να αντιδράσω και το είπα και στον πρόεδρο Φανορομπά, με εξέπληξε η στιγμή που αποφάσισε να μιλήσει για αυτή την ιδέα. Για την ιδέα αυτή, για ένα νέο προπολογισμό, την παραμονή των διαπραγματεύσεων που γίνονται για τον κοινοτικό προπολογισμό, και μάλιστα τη στιγμή που οι σε αυτές φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ λεπτές με δύο κατηγορίες ε, χωρών που αντιτίθεται, γιατί μεν θέλουν να παγώσει, να μειωθεί ο κοινοτικός προπολογισμό, οι άλλες θέλουν να αυξηθεί, καταλαβαίνετε ότι αν μη τι άλλο δεν ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή. Από εκεί και πέρα. Χέλγα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εξετάζοντας την γνωμοδότησή μας που θα σας παρουσιάσω την επόμενη εβδομάδα και ενδεχομένω να εγκρίνουμε και τροπολογίες ή να προτείνουμε τροπολογίες στο κείμενο της κυρίας ε, Τάισεν, την οποία είδα χτες και είναι εντελώ ανοιχτή σε ό,τι θέλουμε εμείς να τις προτείνουμε. Φυσικά θα πρέπει να δούμε την επόμενη εβδομάδα όταν ψηφίσουμε την προσωρινή έκθεση, είτε εμείς στην Επιτροπή μας, είτε στην ολομέλη, είτε ανάμεσα στην επόμενη εβδομάδα και την ολομέλη να δούμε κατά πόσο στο κείμενο της κυρίας Τάισεν ή στο δικό μας κείμενο θα προσθέσουμε μια παράγραφο, κάτι που να αναφέρεται σε τέτοιου είδους ιδέες. Όπως η Χέλγα, έτσι κι εγώ έχω εκπλαγεί και κάπως ανησυχώ που βλέπω να εισάγεται ένα επιπλέον στοιχείο σύγχυσης σε μια συζήτηση που έτσι καλώς είναι δύσκολη. Άλλες παρατηρήσεις παρακαλώ. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε ελεύθεροι. Και δίνουμε ραντεβού για την Δευτέρα στις 3 το απόγευμα, προκειμένου να εξετάσουμε το σχέδιο προσωρινής έκθεσης. Έληξη συνεδρίαση.